Είχε ήδη ενοποιήσει την Ευρώπη, ακόμα και οι τόρις χειροκρότησαν. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση την Επιτροπή για την συζήτηση. Τώρα θα έρθουμε στην ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου. Ε, ο συνάδελφος κ. Κέναν έθεσε ένα αίτημα βάσει του άρθρου 177. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, Σύμφωνα με το κανονισμό 177 για το διαδικαστικό, θα ήθελα να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία για μια περίοδο τριών μηνών. Και ο λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί μια απόφαση για αυτό το θέμα τώρα. Λάβαμε μόνο την απόφαση του δικαστηρίου στι 14 Σεπτεμβρίου και οι περισσότεροι βουλευτέ δεν είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν αυτή την απόφαση κατάλληλα. Γιατί να γίνει εσπεσμένη αυτή η ψηφοφορία. Δεν υπήρξε καμία δυνατότητα να εξεταστεί κατάλληλα η απόφαση του δικαστηρίου και δεν υπήρξε δυνατότητα να υπάρξει νομική γνώμη εν σχέση με το τι ακριβώς σημαίνει από νομική άποψη αυτή η απόφαση. Εσείς κύριε Πρόεδρε αποφασίσατε να μην υπάρξουν τροπολογίες που προτείνουν να υπάρξει αλλαγή όσον αφορά τις ε, τέσσερις μέρες της Συνόδου. Εγώ θα ήθελα να έχετε μια νομική τεκμηρίωση για κάτι τέτοιο. Ε, οι περισσότεροι βουλευτές δεν έχουν δει ακόμα το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν αποσταλεί αντίγραφα, υπάρχει μόνο στην ιστοσελίδα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω γιατί έχει προωθεί με αυτό τόσο σπισμένα. Και τέλος, ε, μια μεγάλη ψηφία στο το σώμα υπερψήφισαν στο να, το να περνάμε λιγότερο χρόνο στο Στρασβούργο εξοικονομώντα ε, βενζίνη, χρόνο και χρήμα, εκπομπέ μάλλον καυσαερίων, χρόνο και χρήμα συμφωνούμε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά ζητάμε για μια λογική ε, μετάθεση. Ε, κύριε Πρόεδρε, να δοθεί δυνατότητα στη διάσκεψη των Προέδρων να αξιολογήσει πάλι αυτή την απόφαση και ίσως να μπορέσει και το Συμβούλιο να, πάρει, ε, να βάλει ένα τέλος σε αυτά τα ταξίδια. Ευχαριστούμε πολύ ο χρόνος αγόρευσης είναι περιορισμένος για τέτοιου είδους αιτήματα, αλλά επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, σας επέτρεψα ε, να μιλήσετε παραπάνω. Είναι κάποιος υπέρ αυτού του αιτήματο, θέλει να μιλήσει υπέρ. Eh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ με αυτές τις ε, θεωρίες συνωμοσίας στις οποίες αναφέρθηκε ο συνάδελφος. Εκπροσωπώντας πάντως τη σουηδική αντιπροσωπεία στη δική μου πολιτική ομάδα, θα ήθελα να σα πω ότι εμεί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να βιαστούμε αυτή τη στιγμή με το ζήτημα του χρονοδιαγράμματο. Ακολουθούμε ήδη ένα χρονοδιάγραμμα, το έχουμε εγκρίνει. Το νέο χρονοδιάγραμμα, αν δεν κάνω λάθο, μέχρι το καλοκαίρι είναι ταυτόσιμο με το υφιστάμενο. Επομένω, δεν τίθεται κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε ενδεχομένω η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων να αναλύσει λίγο περισσότερο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο κατά του αιτήματο αυτού, ο κύριο Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώ να θέσω ένα ερώτημα. Εγώ διάβασα την απόφαση του δικαστηρίου και συνήθω το χρονοδιάγραμμα για το 2013 έχει ακυρωθεί το χρονοδιάγραμμα και καθώ έχει ακυρωθεί το χρονοδιάγραμμα ακούγοντας συναδέλφου, αυτό σημαίνει ότι από τη Δευτέρα δεν θα μπορέσουμε να συνεδριάσουμε πουθενά ούτε καν στις Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν θα έχουμε διακοπέ. Αυτό θα μα δώσει λοιπόν τρει μήνε προβληματισμού εν σχέση με το πώ θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα για το 2013. Ευχαριστώ πολύ. Άρα η πρόταση βάσει του άρθρου 177 παράγραφος 2 είναι υπέρ της αναβολής. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής. Ποιος είναι κατά. Απέχει. Άρα δεν γίνεται δεκτό. Ευχαριστώ πολύ. Απορρίπτεται. Και τώρα θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν. Θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση της πρότασης του κ. Κιάνεν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα θα περάσουμε στη ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Είναι, έχει αρκετή ζέστη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη ψηφοφορία. Καταρχήν, έλαβα από το EFT ε, το αίτημα να διοριστεί ο κύριος Μπέλντερ ε, ως μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ιαπωνία στη θέση του, του Μάικ Νάτρασα σύμφωνα με το κανονισμό 164 παράγραφο 2 δεν υπάρχει αίτημα να ψηφιστεί το